Θα ήθελα να ζητήσω από τους συντάκτες της ε, έκθεσης να πάρουν το λόγο. Κυρία Σοπράνη. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο νέος της Αλήμ Εμρ ε, καταδικάστηκε σε θάνατο ε, στην ε, Σαουδική Αραβία ενώ ήταν μόλις 17 ετών την εποχή εκείνη που υποτίθεται ότι συμμετείχε σε διαδηλώσεις αντιπολιτευόμενων στους ΣΥΙΤΕΣ. Δεν έχει κάνει ποτέ, ποτέ κανένα έγκλημα. Τα δικαιώματά του για μια δίκαιη δίκη ποτέ δεν είναι γίνει σεβαστά. Η περίπτωση αυτού του νέου ΣΥΙΤΗ μας επέτρεψε να βρούμε στις ομάδες μεγάλη συνένεση και χαίρομαι γι' αυτό. Ε, ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, των υπολείπων ομάδων. Ε, έχουμε ένα κείμενο το οποίο δεν χαρακτηρίζεται από τη βούληση να καταδικάσουμε μια ολόκληρη χώρα, αλλά να τη λογικεύσουμε όσον αφορά κάποιε πρακτικέ, οποίες, οι οποίες δεν είναι πλέον αποδεικτέ όταν θέλουμε να ανήκουμε στην κοινότητα των εθνών. Ε, ε, οι Σαουδάραβες καταναλώνουν ε, την υψηλή μας τεχνολογία, αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να δικαιολογήσουν αυτά, αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος ο κύριος και Είναι τραγική ηρωνία ότι τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία υποτίθεται θα είναι επικεφαλής ε, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, σε μια σημαντική επιτροπή καταδικάζει έναν ε, έφηβο για μόνο το έγκλημα είναι ότι διαμαρτυρήθηκε, συμμετείχε στη διαμαρτυρία. Όμως χτες μόλις προέκυψαν και άλλες εκθέσεις για τον Ταούντα Αλμαχούρ που αντιμετωπίζει την ίδια μοίρα έχει, βρίσκεται στη φυλακή από το 2012, είναι μόλις 17 ετών ο Λίμα ε, ε, Νέμρ. Ε, δεν είναι μόνο έγκλημα, αλλά είναι γενικά ένας ευρύτερος πόλεμος της Σαουδικής Αραβίας ενάντια σε συγκεκριμένης προέλευσης ε, ε, ανθρώπους, ε, τους ήτες Αυτές είναι πολύ σοκαριστικές υποθέσεις, αλλά υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος κατάχρησης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία. Γιατί είναι ένα καταπιεστικό και αυταρχικό κράτος. Καλούμε τη Σαουδική Αραβία να δώσει χάρη στον Αλνίμερ καθώς και στον Αλ Η κυρία Ρίς. Ναι, εκείνος είναι, έχει 17 ετών. Ένα παιδί ένα παιδί, ένας φοιτητής ε, πρότυπο που του αρέσει η φωτογραφία, το ποδήλατο, του αρέσει η ελευθερία και από ό,τι φαίνεται του αρέσουν και τα πόλο Ραλφ Λόρεν, τα μπλουζάκια Ραλφ Λόρεν. Όπως πολλοί χιλιάδες άνθρωποι στους οποίους είχε δώσει φτερά η Αραβική Άνοιξη ε, στην ε, δεν έγινε αραβική άνοιξη εκεί για τον Αλή ε, τον ε, ε, βούτυξαν, τον συνέλαβαν τέσσερα χρόνια βρίσκεται στη φυλακή εδώ βλέπουμε τον Αλή, το οποίο έκλεψαν την νεότητα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί σε θάνατο, μπορεί αύριο μεθαύριο να εκτελεστεί η ποινή αυτή. δεν επανέρχομαι στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σαουδική Αριβία. το κάνει το κείμενό μας η Σαουδική Αραβία τοποθέτησε στο υψηλότερο επίπεδο τώρα το πρέσβη της στα Ηνωμένα Έθνη. Ζητώ χάρη για τον Αλή Αλνίμρ. Ο κύριος Κοράου τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Σαουδική Αραβία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάλι για το ίδιο θέμα μιλάμε. Τεράστια συνέπεια στη στάση μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Σαουδική Αραβία που τη θεωρούμε τα έρωμα μας ε, ε, μια χώρα με την οποία διατηρούμε καλές σχέσεις, μια χώρα που δεν πρέπει να την καταδικάζουμε, είναι μια από τις χώρες στον κόσμο όπου γίνονται οι χειρότερες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όπου θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο αυστηροί. Αντίθετα τι συμβαίνει για να καταδικάζουν ε, σε σταύρωση ή σε θάνατο με όλους τους πιο φρικαλαίους τρόπους, εμείς τους επιβραβεύουμε και τον βάζουμε και τον δικό τους ε, επικεφαλής ε, της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον ΟΗΕ, άκουσαν, άκουσαν, με υποστήριξη των Βρετανών. Ο Κάμερον δεν ήξερε τι να πει. Ε, ε, όταν το ρωτήσαμε. Το στηρίζουμε λοιπόν ε, συστηματικά. Μα συνάδελφοι, τι είδου προσέγγιση είναι αυτή απέναντι στην Σαουδική Αραβία. Πρέπει να μάθουμε να την καταδικάζουμε και να, την, και να τις επιβάλλουμε ποινές. Γιατί φορτικά καλύτερα να πάψουμε να μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Αλή Αλνίμρ συνελήφθηκε, βασανίστηκε επειδή συμμετείχε στην Αραβική Άνοιξη. Δεν πρέπει να ε, αφήσουμε να τον θανατώσουν. Έχει να αντιμετωπίσει ένα φρικτό θάνατο. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι πρώτον ότι δεν θα εκτελεστεί και δεύτερον ότι θα μπορεί να επιτρέπονται ειρηνικές διαδηλώσεις Σαουδική Αραβία η οποία παραβιάζει ε, τις υποχρεώσεις ε, που επέχει λόγω του ότι είναι συμβαλόμενο μέρος σε Σύμβαση ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών. Ίσως επειδή είναι από οικογένειες ητών και αντιφρονούντων είναι σε αυτή τη δινή θέση ο Αλή Αλνίμρ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε ότι θα πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα η Σαουδική Αραβία. Το παιδί αυτό ε, καταδικάστηκε σε θάνατο ως τρομοκράτης όμως φαίνεται να εξαναγκάστηκε να ομολογήσει μετά από βασανιστήρια και σε μια δίκη που έγινε μυστικά. Πραγματικά ε, μου προκαλεί ε, αποτροπιασμό το γεγονός ε, ότι βάζουμε και η χώρα μου πρωτοστατεί έναν άνθρωπο από αυτή τη χώρα στην κορυφή ενός οργανισμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτά που καταπατάει η χώρα. Υπάρχουν υποσχέσεις ε, που έχουν δοθεί και αν σημαίνουν κάτι θα πρέπει αυτό το πεδίο αλή να ζήσει για να γίνει άντρας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεχόφσκι, επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε. Το κείμενο αυτό ε, καταδεικνύει ακόμη μία παραβίαση ανθρωπινών δικαιωμάτων ε, στη Σαουδική Αραβία. καλό είναι να έχουμε και οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Πολύ σημαντικό όμως είναι να διατρανώσουμε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ο Αλή Μοχάμετ Αλνίμερο παραβιάζεται ε, με την περίπτωση ε, της ε, καταδίκης του σε εκτέλεση η Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και η Αραβική Χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. όλοι οι αξίες μας καταπατώνται με αυτή την καταδίκη. Από το 2014 ο αριθμός ε, των ε, θεατικών ποινών αυξάνεται στη Σαουδική Δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια προς αυτήν την κατάσταση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ε, σα ευχαριστώ κυρία Βερζιά. Έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ο ρόλος αδική ε, Αραβίας που είναι ένας αποσταθεροποιητικός ρόλος φαίνεται και στην Ιεμένη αλλά και με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. Αλλά βλέπουμε τον πανικό και το, το, την τρομοκρατία και μέσα στην ίδια τη χώρα διακριτική μεταχείριση, κακοποίηση ε, γυναικών ε, ζει ε, πραγματικά στο μεσαίο ακόμη χώρα. Βλέπουμε τις φωτογραφίες του Αλή Αλνίμερ, θύμα μιας άδικης δίκης, βασανισμένος, κακοποιημένος ο οποίος απλά τι έκανε, διαδήλωσε μόνο για τα δικαιώματα του λαού του και το λάθος του ήταν ότι ήταν ανυψιός ενός αντιφρονούντα. Αυτοί που πρέπει να δράσουν όμω ε, κοιτάνε αλλού και αφήνουν να λαμβάνει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ Σαουδική Αραφία και η Γαλλία, η Βρετανία. Είναι καλύτερη σύμμαχοι. Δεν θα πρέπει να ε, πεθάνει ο Αλή Αλνίμρα. Ούτε όμω και ο άλλο νερό που συνελήφθη θα πρέπει ε, να. ο, θα πρέπει να υποβληθεί σε μαστίγωση. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένας νέος 20 ετών ε, που κινδυνεύει να δολοφονηθεί λόγω της, ε, του κινησμού και της αδιαφορίας. Ο κινησμός μιας δικτατορίας ε, που υπογράφει ένα σωρό συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών ε, για να, ε, και συνεχίζει διαφορετικά να, να λειτουργεί. Η διαφορία είναι αυτών που συνεργάζονται με μια τέτοια κυβέρνηση για να, πουλών, για, για να μπορούν να παίρνουν πετρέλαιο και για να πουλάνε όπλα. Ας μην αφήσουμε την Ευρώπη να θυσιάσει τις αξίες της ε, για ένα ξενοδοχείο, να μπορεί να μένει σε ένα ξενοδοχείο μιας αιματοβαμμένης δικτατορίας. Δεν σκοτώνουμε ένα παιδί, δεν το καταδικάζουμε σε θάνατο. Και ναι, ζητήσαμε τη χάρη, αλλά πέρα από αυτό πρέπει να ζητήσουμε από την Σαουδική Αραβία να φτιάξει μια επιτροπή έρευνα κατά των βασανιστήριων και έτσι ώστε οι ατομικέ ελευθερίε και τα ανθρώπινα δικαιώματα να γίνονται σεβαστά σε αυτή τη χώρα. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ο κύριος Πόσπης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με όλους αυτούς τους ομιλητές που καταδίκασαν τις, ε, τη βαρβαρική εκτέλεση που προγραμματίζεται του νέου αυτού. Και στον 21ο αιώνα η τιμωρία δεν μπορεί να έχει αυτή τη μορφή. Δεν είναι δυνατόν να σταυρώνουν και να αφήνουν το σώμα του ανθρώπου να σαπίζει στο σταυρό για την έκφραση πολιτικών ιδεολογιών, για το γεγονός ότι είναι Σιήτης, για το γεγονός ότι είναι ανιψιός του θείου του, ένας αντιφρονούντας ε, με μεγάλη επιρροή στη Σαουδική Αραβία. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ως ε, ίσο εταίρο την Σαουδική Αραβία. Δεν μπορούμε να αποστρέψουμε το βλέμμα μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει αυξηθεί δυστυχώ ο αριθμό των εκτελέσεων. 102 οι εκτελέσεις ε, φέτος και συνεχίζονται οι παιδιά, ξένοι. Εκτελούνται χωρίς εγγύηση δίκαιης δίκη. Τρίτη είναι στον κόσμο η Σαουδική Αραβία στον αριθμό των εκτελέσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος και τώρα δίνει το λόγο στην κυρία Γκόμες. Όλη η Μουχαμέταλ έχει καταδικαστεί σε θάνατο με αποκεφαλισμό και μετά επιπλέον σταύρωση. Μεσαιωνική τιμωρία, βία, ε, ε, διώκονται ε, ε, λόγω της ε, ελεύθερης έκφρασης και επειδή δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα. Η ύπατη εκπρόσωπος, η Φρεντερίκα Μογερίνη, θα πρέπει δημόσια να εκφράσει τη φρίκη μας για αυτή την καταδίκη που πλήττει τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να γίνουν όλες οι προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα για να τεθεί τέλος στη βαρβαρία. Αν σκεφτούμε ένα σωρό άλλες περιπτώσεις όπως ε, η μαστίγωση του Γαΐθ Μακτάου, ε, θα πρέπει να επανεκτιμήσουμε με βάση όλα αυτά τις σχέσεις που έχουμε με την ε, Σαουδική Αραβία. Εμπόριο, συνεργασία, στρατιωτική. Είναι αβάσταχτη η σιωπή των ευρωπαϊκών χωρών. Ανταλλάσσουν πετρέλαιο με όπλα. Είμαστε συνένοχοι εφόσον σιωπούμε. Ο Πρόεδρος Διακόπτη. Ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Δεμεσμάκαρ. Σας ευχαριστώ. Ένας νεαρός 17, 17 ετών συλλήφθηκε, ε, βασανίστηκε και τώρα καταδικάστηκε σε θάνατο αποσταύρωση. Τέτοιες ε, πρακτικές, εγώ το συνδέω με την, ε, το Ισλαμικό κράτος, με την Αλικάιντα. Η Σαουδική Αραβία έχει επενδύσει εκατομμύρια στην ε, καταπολέμηση της πολιτισμικής μουσουλμανικής κοινότητας και σήμερα όλοι αυτοί είναι υπό την ηγεμονία του Σαουδικού Βαχαμπισμού και είναι κατά της Δύσης, κατά της ε, σύγχρονης ε, εξέλιξης, κατά των δικαιωμάτων των γυναικών. Και η συνέλευσή μας πάντα ήταν πολύ αυστηρή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισοδική Αραβία. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι εξαγοράζονται πολύ εύκολα από τα πετροδόλαρα ή κάποιοι ηγέτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη σε ό,τι αφορά τον Άλλη Μοχάμετα Θα πρέπει να δοθεί ε, άφεση. Uh, Madam Chair, uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κυρία Πρόεδρε, ακούσαμε ότι είναι σημαντική χώρα στη Μεσανατολή Σαουδική Αραβία και πιστεύω ότι έχουμε κοινού στόχου ε, για την ειρηνευτική διαδικασία. Και φυσικά θα πρέπει να κοιτάξουμε από κοινού κάποια ζητήματα. Είναι κοινό συμφέρον μας αυτός σωστά αναφέρθηκε ότι το ιστορικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα της αντιξαραβίας είναι τραγικό. Και νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε λοιπόν άλλη μια τέτοια περίπτωση σε ό,τι αφορά αυτό το ιστορικό. Και θα πρέπει να επαναλάβω αυτά που είπε ο, ο πρόεδρος Ολάντ. Μίλησε εξ ονόματο μιας χώρας με παραδοσιακού ισχυρού δεσμού με την Σαουδική Αραβία. Έκανε λοιπόν μια ισχυρή δήλωση προ την Σαουδική Αραβία. Αυτό που μα λείπει είναι μια σαφή τοποθέτηση τη κυρία Μογκερίνη. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι εδώ αναμένουμε να δείξει σκληρή γραμμή η κυρία Μογκερίνη και θα πρέπει να συμφωνήσουμε αν συνεχίσει αυτή η πορεία θα πρέπει να υπάρξει μια ηχηρή και στεναρή αντίδραση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα κοινά ζητήματα και τα κοινά συμφέροντα που έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ελέη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, όπως και όλοι εδώ νομίζω ε, δεν μπορούμε να αρκούμε σε αυτές τις ε, τυπικές ε, διαμαρτυρίες. Κάθε θεσμικό όργανο της Ένωση πρέπει να κάνει πάντα το δυνατό για να αποτραπεί αποκεφαλισμός και η σταύρωση του Αλ Νίμερ. Πάνω από 2.500 εκτελέσχαμε τα τελευταία χρόνια. Η Σαουδική ε, Αραβία ε, είναι στην Άβυσσο, στη βαρβαρότητα μιας άλλης εποχής, ε, ζει στο Μεσαίωνα. Δεν μπορούμε να δείξουμε καμία αυταρέσκεια. Θα πρέπει και να ακουστεί φωνή μας ε, πιο ηχηρή και να αναλάβουμε δράση. Ακόμη και αν τεθούν υπό αμφισβήτηση κάποιε συμφωνίε εμπορικέ κτλ. Γιατί τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη αξία από την ανθρώπινη ζωή. θα πρέπει η Προεδρία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, ε, των Ηνωμένων Εθνών ε, να μην δοθεί στη Σαουδική Αραβία. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους δύο νέους, τον Αλνίμρα και τον Ελμαρούν. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Βαλενθιάν. Η Σαουδική Αραβία θα αποκεφαλίσει ένα νερό που ε, διάπραξε ένα δίκαιο μα ηλικία 17 ετών. Έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ ε, η Σαουδική Αραβία, η δικαιοσύνη της. 130 άτομα έχουν αποκεφαλιστεί φέτος και αυτό, ε, αυτή τη φρικτή μοίρα περιμένει και τον Αλή εάν εμείς δεν υψώσουμε τη φωνή μας πέρα της απελευθέρωσής του. Το Κοινοβούλιο δεν θα πάψει να αναφέρει ε, πόσο απάνθρεπη είναι η δράση της κυβέρνησης και της δικαιοσύνη. Οκτώ μήνες μετά την έγκριση κατεπήγοντος για την ε, περίπτωση του Γαΐθ ε, που ζητούμε να απελευθερωθεί και σήμερα, το Κοινοβούλιο θα ψώσει τη φωνή του σήμερα και για τον Αλή Αλνίμρα. Δεν πρόκειται να σιωπήσουμε. Η Σαουδική Αραβία, η κυβέρνηση πρέπει να το καταλάβει. Δεν μπορεί να αποκεφαλίζει αθώους νέους ανθρώπους που το μόνο έγκλημα που έκαναν ήταν να αγωνιστούν για την ελευθερία τους. Σας ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνεται και αυτός ο γύρος και δεν υπάρχει διαδικασία catch the eye που να προβλέπατε και δίνει το λόγο λοιπόν στον κύριο Στελιανίδη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι αξιότιμοι βουλευτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θέτετε την περίπτωση του κυρίου Αλή Μοχάμετ Αλήμρ. Όπως γνωρίζουμε, η Σαουδική Αραβία αποτελεί σημαντικό εταίρο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά, όπως ε, πολλοί στην Ευρώπη, και εμείς ε, ανησυχούμε από την καταδίκη σε θάνατο στον, ε, που επιβλήθηκε στον Άλλη Μοχάμετ Αλήμρ στις αρχές του έτου. Ήταν ανήλικος όταν συνελήφθη το 2012 μεταξύ άλλων για τη συμμετοχή σε εγκληματικές ομάδε και μετά από συμμετοχή σε διαμαρτυρίε ε, στην ανατολικέ Επαρχίες και παρακολουθήσαμε τι εξελίξει σε ό,τι αφορά την υπόθεση του καθώ και την γενικότερη κατάσταση σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Σαουδική Αραβία η βάση και οι όροι ε, τη καταδίκη ε, του κυρίου Άλλη Μοχάμενταν Ρήμ καθώς και η φύση της τιμωρίας της ποινής αποτελούν ζητήματα που ανησυχούν εντονότατα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η ποινή φαίνεται ε, εξόφθαλμα δυσανάλογη. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σε στενές, επαφές ε, με τις ε, αρχές του Ριάντ και μας ζητήθηκε να διαβιβάσουμε την έντονη αντίληψή μας για την δυσαναλογία της ποινή και να απευθύνουμε έκκληση στις αρχές της Αντικής Αραβίας να επαναεξετάσουν την ποινή και την καταδίκη του κυρίου Αλή Μοχάμεντ Ιρέμπρε. Και αυτό αφορά ασφαλώ και την θέση επί τη αρχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη θανατική ποινή, καθώ και την ανησυχία τη επιβολή τη θανατική ποινή στην Σαουδική Αραβία. σε σεβασμού των ελάχιστων προτύπων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θέματα της εκτέλεσης ανηλίκων, καθώς και να δώσουμε μια χείρα για να δώσουμε χείρα βοηθείας και να μπορέσει να υπάρξει μια συζήτηση. Πραγματικά φτάνει σε επίπεδα άνευ προηγουμένου η θανατική πίνη στην Σαουδική Αραβία. Ε, τέτοιες ποινές επιβάλλονται ακόμα και για ε, εγκλήματα, για αδικήματα που έχουν να κάνουν με τα ναρκωτικά, για παράδειγμα. Άρα ζητούμε από την Σαουδική Αραβία να επανεξετάσει την ε, ποινή του κυρίου Άλλη Μοχάμετ Ανδρέη Σας διαβεβαιώνουμε λοιπόν ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή και να ανακοινώνουμε ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Επιτροπέ Λέγη Πρόεδρε, για τα καταλητικά αυτά σχόλια και θα ήθελα να στήσω συγγνώμη για τον θόρυβο που επικρατεί στην αίθουσα της Ολομέλειας, αλλά βλέπετε έχουμε και 751 μέλη, 751 βουλευτές. Ε, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο το επίπεδο του θορύβου και γι' αυτό σας ζητώ συγγνώμη. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ζητήσω στο σημείο αυτό να καθίσετε και όσοι εισέρχεστε στην αίθουσα παρακαλώ να εισέρχεστε προσεκτικά και χωρίς θόρυβο. Έχουμε οκτώ ψηφίσματα, σχέδια ψηφίσματο ε, που έχουν κατατεθεί και ολοκληρώνεται λοιπόν στο σημείο αυτό η συζήτηση και σε λίγο θα ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. So, colleagues, I ask everybody to sit. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε όλοι για να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες, ε, διαδικαστικό, κυρία Ζώμη. Um Έχω ένα διαδικαστικό, κυρία Ζούμπερ, σύμφωνα με το 130 άρθρο του κανονισμού. το να υπάρχει ανώτατο όριο για υποβολή γραπτών ερωτήσεων για κάθε βουλευτή είναι κάτι το φρικτό. Εμείς πρέπει να δικαιολογήσουμε ότι είναι επίγον το αίτημά μας και το ερώτημά μου. Εχθές μάλιστα έλαβα μια απάντηση από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου που απέρριψαν μια ερώτηση που επέβαλα γιατί δεν το θεωρούν επίγον να τον ρωτήσω ε, τον Επίτροπο για το τι γίνεται με τις αστυνομικές, ε, μάλλον στρατιωτικές δυνάμεις και τους πρόσφυγες τι ε, τις τελευταίες ημέρες. Πώς γίνεται ένας γραφειοκράτης να αποφασίζει αν είναι επίγουσα πήγουσα η ερώτησή μου. Οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου εξυπηρετούν την εργασία των Ευρωβουλευτών ή να θέλουν να την παρεμποδίζουν. Δεν κατάλαβα. Συνάδελφε Ζούμπερ, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω όμως ότι δεν πρόκειται για γραφειοκράτες αλλά για την ολομέλεια του Κοινοβουλίου που στην τελευταία σύνοδο αποφάσισε να περιορίσει τον αριθμό των γραπτών ερωτήσεων. Λυπούμε, αυτό είναι ένα γεγονός, είναι μια πραγματικότητα, η ολομέλεια αποφάσισε πάνω σε αυτό. Και τώρα ερχόμαστε στις ψηφοφορίες. Να πω ότι τα πρακτικά της θεσινής συνόδου είναι διαθέσιμα, υπάρχουν σχόλια. Όχι.